Good Καλημέρα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε την σημερινή μερίσια διάταξη. Δεν έχει κανείς ε, καμία αντίρρηση, οπότε εγκρίνεται. Σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίαση αυτή, την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και περιβάλλοντος ε, για το τρίτο αυτό πακέτο της ε, ταξινόμησης έχουμε και τους άλλους δύο φακέλους για την αποκαλύψη, την αποκάλυψη και τη συγκριτική αξιολόγηση ε, που συνεχίζονται. Είχαμε τις πρώτες τριμερείς διαλόγους την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και επίσης είχαμε και μια συνάντηση για αυτό εδώ το θέμα και χαίρομαι που υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των συνεισηγητών που θα μας ε, βοηθήσει να επιτύχουμε μια ε, ισχυρότερη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε συνεδρίαση για μία ώρα. γιατί έχουμε προγραμματίσει και ψηφοφορία μετά, μέσω μετά τη συζήτηση. Οπότε... Θα ήθελα να δώσω αμέσω ε, τον λόγο στους δύο συνεισηγητές για έξι λεπτά στον ε, καθένα. Δίνω τον λόγο πρώτα απ' όλα στην ε, κυρία Πιετικάινεν. Παρ' όλα αυτά, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Μπας Άικχαουτ, ε, τον συνεισηγητή μου και τα άλλα μέλη της Επιτροπής που συνεισέφεραν σε αυτήν την έκθεση και τις προηγούμενες εκθέσεις ε, για τη συγκριτική αξιολόγηση, την έκθεση ιδίας ε, πρωτοβουλίας και την αποκάλυψη. Βεβαίως πρόκειται για ένα ευρύτερο πακέτο για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, πως οι δείκτες αυτή βιωσιμότητας ε, και η συνοχή ακριβώς θα προωθηθεί στον τομέα αυτόν. Και βεβαίως ε, η συνοχή εδώ πέρα είναι το σημαντικότερο τμήμα γιατί διαφορετικά στέλνουμε παραπλανητικά μηνύματα. Και έχουμε διαφορετικές απαιτήσει από διαφορετικούς κλάδους ε, επενδύσεων και αυτό το οποίο συμφωνήσαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων ε, και στις δύο είναι ακριβώ να διατηρηθεί η σύνδεση και η συνοχή μεταξύ των δύο εκθέσεων και θέλω να το αναφέρω αυτό πρώτα απ' όλα στην αρχή γιατί εξηγεί τις αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την έκθεση. Οπότε, το ερώτημα είναι το Έχουμε αλλάξει το πεδίο εφαρμογή σε όλους του συμμετέχοντες αντί να καθορίζουμε μόνο το ποιοι ακριβώς καλύπτονται. Γιατί αν αρχίσουμε να τους καθορίζουμε το πρόβλημα είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε φούσκε. Δεύτερον είναι πάντα δύσκολο να τους καθορίσουμε επακριβώς και τρίτον βεβαίως υπάρχει το θέμα του αντικτύπου στο κλίμα και άλλου από κλάδους όπως ο κατασκευαστικός δεν μπορούμε να πούμε ότι το μπετόν είναι φιλικό προς ε, το περιβάλλον ε, και να μιλήσουμε για πράσινες επενδύσεις. Οπότε στόχος είναι να δώσουμε τις πληροφορίες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά για τον αντίκτυπο που έχουν ε, οι διάφορες ε, δραστηριότητες σε όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος, δηλαδή την κατανάλωση πόρων, ε, την επίδραση στη βιοπικιλότητα, στις εκπομπές, στη χρήση γης και βεβαίως στη χρήση του νερού και βεβαίως στην κλιματική αλλαγή. Μετά. περιβαλλοντική λογιστική θα λέγαμε και εκεί πέρα μπορούν να δοθούν περισσότερες οφορίες και να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην αγορά να καθορίσει σε ποια φάση του μετασχηματισμού βρίσκονται οι διάφορες εταιρείε ε, εντό ενός κλάδου. Κάτι άλλο το οποίο προκύπτει από αυτό το σκεπτικό είναι το πεδίο για να καλυφθούν όλοι οι συμμετέχοντες στις ε, χρηματαγορές όχι μόνο όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά όλοι οι δρόντες, τα πιστοτικά ιδρύματα σε αυτήν την φάση περιλαμβάνονται. Τέλος, ε, για το κλίμα, αν δείτε την αρχική πρόταση και τις ε, στρεβλώσεις, ε, ε, η βιοενέργεια είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά μπορούμε να δούμε παραδείγματος χάρη το παράδειγμα του φινικελαίου. Δηλαδή από την πλευρά του κλίματος φαίνεται μια καλή επένδυση, αλλά αν δούμε τον συνελικό αντίκτυπο, παραδείγματος χάρη στο περιβάλλον, στη βιοπικιλότητα δηλαδή, η, την χρήση των δασών, τότε είναι τελείως αρνητικός ο αντίκτυπος. Μετά, οι κοινωνικές ε, πτυχές και οι πτυχές της διοίκησης ε, επίσης περιλαμβάνονται. Το θέμα είναι βεβαίως το πόσο μακριά θα πάμε αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ζήτημα ε, πολιτικής συζήτησης. Βεβαίω, ε, όλα αυτά θα τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρότερη εποπτεία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και θα πρέπει ίσως να δοθούν περισσότερες ή ισχυρότερες αρμοδιότητες στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, γιατί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι ο ίδιος, γνωρίζουμε πρώτον και δεύτερον βεβαίως μιλάμε για εσωτερική αγορά και χρειάζεται ίση ώρα ανταγωνισμού για όλους τους δρόντες. Και βεβαίως τα βασικά στοιχεία της κατάταξης το σκεπτικό εδώ είναι να ορίσουμε τους κανόνες για τους ε, δείκτες, ε, δηλαδή Ποιο περιβαλλοντικό αντίκτυπος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ναι, και υπάρχουν διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει. Τίποτα το πολύ δραστικό όταν μιλάμε για το συνολικό περιεχόμενο, αλλά για την βιοπικιλότητα. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν μετά κάποιες ανάγκες να δούμε π.χ. την σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, αναφέρω τα LULUCF παραδείγματο χάρη, γιατί βεβαίω αυτά είναι ζητήματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. και πρέπει να ληφθούν, όταν θα εφαρμοστεί, να ληφθούν υπόψη όταν θα εφαρμοστεί ο κανονισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι γενικά τα σημεία. Υπάρχουν κάποιες ε, πολύ καλές ε, τροπολογίες ε, και Ήδη νομίζω αναφέρθηκε το ότι αναζητούμε κάποιες, ε, κάποιους συμβιβασμούς. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί η η κυρία Πιετικάινεν αναφέρθηκε στα περισσότερα σημεία που συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν πάνω από 500 τροπολογίες για τον φάκελο αυτό από δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οπότε πάλι καλά. Σε άλλα θέματα είχαμε ακόμα περισσότερες τροπολογίες. Αυτό βέβαια δείχνει ότι γενικά πιστεύουμε οι διάφορες πολιτικές ομάδες ότι λίγο πολύ συμφωνούμε με τις επιλογές των συνεισηγητών στο σχέδιο έκθεσης. Φυσικά θα υπάρξουν συζητήσεις. Η κυρία Πιέτη Είχαμε την πρώτη συνάντηση στο Στρασβούργο, οι σκιώδρες εισηγητές, αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για τα διάφορα ζητήματα. Και είναι σαφές ότι χρειάζονται και άλλες συζητήσεις ακόμα. Τα κομβικά στοιχεία είναι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, όπου οι συνεισηγητές λένε ότι αν θέλουμε να προσδιορίσουμε το τι είναι βιώσιμο, πρέπει να προσδιορίσουμε και τι δεν είναι βιώσιμο. Οπότε αυτό το συζητάμε με τους σκιώδεις, οι οποίοι συμφωνούν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει βέβαια να επιλέξουμε και την διατύπωση. Οι περισσότερες τώρα τροπολογίες θέλουν να επεκταθεί η ταξινόμηση και στον κοινωνικό τομέα. Κάτι το οποίο στηρίζουμε μεν, αλλά το θέμα είναι σε τι βαθμό, πόσο μακριά θα πάμε κάτι το οποίο σίγουρα θα μας οδηγήσει σε επιπλέον συζητήσεις. Ε, πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουμε. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε το φάκελο αυτό, το θέμα αυτό, με άλλα ζητήματα ε, τα οποία εξετάζουμε στην κατηγορία βιώσιμα οικονομικά. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τους άλλους φακέλους. Αυτά θα είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, πιστεύουμε ότι σε πολλά ζητήματα μπορούμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβασμούς. Και περιμένουμε να είναι καρποφόρε οι συζητήσεις και να είμαστε έτοιμοι γρήγορα και σίγουρα το Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο πριν σταματήσουμε για τις ευρωεκλογέ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Τώρα, οι εισηγητές. Η πρώτη που έχω στον καταλογό μου είναι η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του εισηγητές Πιτικάνεν και Έκχαουτ. Υπογράμμισαν τη σημασία του φακέλου αυτού. Σας ευχαριστώ για την ενδελεχή ανάλυση, τη λεπτομερή παρουσίαση τη υποβληθή αστροπολογία. Είμαι λακωνική σήμερα. Κατευθείαν στο, στην ουσία. Για 20 Φεβρουαρίου προβλέπεται η ψηφοφορία και θα πρέπει να προτείνουμε στην Ολομέλεια ένα ρεαλιστικό κείμενο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να είμαστε και άκρο φιλόδοξοι. Και μεταξύ των σχεδίων εκθέσεων και των διαφόρων τροπολογιών που προβλήθηκαν από διάφορου συναδέλφου, έχω μόνο τα στατικά για να πετύχουμε τη σωστή συνταγή. Οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε υποστηρίζουν ένθερμα την βιώσιμη οικονομία στην Ευρώπη και στον κανονισμό βλέπουμε ότι είναι βασικό εργαλείο να το πετύχουμε αυτό. Χρειάζεται να διευκολύνουμε τη ροή των οικονομικών ροών προ δραστηριότητε οικονομικέ που είναι βιώσιμε και που επιτρέπουν να συμβάλλουμε αποφασιστικά, όπω υπόθηκε από του συναδέλφου, στη μάχη κατά τη αλλαγή του κλίματο και να έχουμε και ένα μοντέλο αναπτυξιακό που είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την εκμετάλλευση των πόρων. Το Κοινοβούλιο δεν ξεκινά εκ του μηδενός, σε αυτή τη δουλειά και μπορεί να καθορίσει τη θέση του αναπτύσσοντας αυτά που εγκρίναμε ήδη στο ψήφισμα για τη βιώσιμη οικονομία και πιο πρόσφατα στον κανονισμούς που αφορούν την αποκάλυψη της, το disclosure και το benchmarks. Να φωτίσω κάποια σημεία που θεωρώ κεντρική σημασία και που, στα οποία αναφέρονται οι τροπολογίε οι δικέ μου και των συναδέλφων τη ομάδα μου. Η πρόκληση να συνοδεύσουμε αυτή τη μετάβαση που αιτείται προσπάθειε είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε προσέγγιση ε, που καλύπτει όλε τι πτυχέ Εν αυτή τη ενία, όσον αφορά τον αντίκτυπο στον βιωσιμότητα, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε συνολικά την οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επενδύσεων και χρηματοδοτήσεως. Δεν θέλουμε να κάνουμε αξιολογήσει ε, με βαθμολόγηση, αλλά έχουμε σίγουρε πληροφορίε όσον αφορά τη βιωσιμότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων. Έτσι θα μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν ε, ε, ενημερωμένοι τις αποφάσεις και να μπορούν να κινούνται προς περισσότερα, σε καλύτερα επίπεδα βιωσιμότητας ε, λαμβάνοντα υπόψη τι τεχνολογικέ εξελίξει των τομέων. Για να κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα βασικό στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε δείκτε. Αυτό ήδη αναφέρθηκε. Δεν θέλω να το επαναλάβω κι εγώ. Θέλουμε δείκτε που εν μέρει ήδη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από την χρηματοπιστωτική αγορά, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ενδεχομένω για ομοιογενή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δείκτε αυτοί που προτείνουμε θα πρέπει να εντοπιστούν και να αναπτυχθούν στις κατεξοδότηση, μέσω κατεξοδότησης ε, πράξεων. Χρειάζεται να το αναλύσουν αυτό οι διάφορε ομάδες των επιτροπών και χρειάζεται να έχουμε μια βάση ευαισιμότητα στην ανάπτυξη και γι' αυτό χρειάζεται σωστή διαβούλευση με του εκπροσώπους των διαφόρων κατασκευαστικών τομέων και από την αρχή να συμμετάσχουν σε αλλαγές που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να εμπλακούν αυτοί οι φορείς ε, άμεσα. Πρέπει να διευρύνουμε και το πεδίο εφαρμογή και να καλύψουμε όλες τι οικονομικές δραστηριότητε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ο τομέας, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες των τομέων, αλλά και τον, κύκλο, τον τρόπο παραγωγής και τον κύκλο ζωής των προϊόντων να επαναλάβουμε και εν ονόματι και τη συναδέλφου Ένελα Τζεντήλε που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα ότι είναι σημαντικό για την ομάδα μας ήδη στον κανονισμό να λάβουμε υπόψη τις τρεις διαστάσεις βιωσιμότητας, δηλαδή περιβαλλοντική πτυχή, κοινωνική και οικονομική διακυβέρνηση. Να συνοδεύσουμε αυτή εξ αρχή του περιβαλλοντικού στόχου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα νέο στόχο που θα έχει στόχο την οικονομική δραστηριότητα ε, του κοινωνικού τομέα. Η πρόκληση για τη βιωσιμότητα συναθρίζει το περιβάλλον και την κοινωνική ένταξη και αυτός ο κανονισμός θα πρέπει αυτό να το αναγνωρίζει ρητά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βιαρίνκ. Αγαπητοί συνεισηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι θέλετε και συμφωνώ επί της αρχής. Έναν ιδανικό κόσμο, όλοι οι επενδυτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές συγχρόνω. Εγώ γνωρίζω τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, ε, δημιουργεί αίσθηση. Και εδώ βρισκόμαστε για να αποφασίζουμε ρεαλιστικά και με λογική και όχι συναισθηματικά τι θέλουμε για το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μια καλή ισορροπία γιατί προσφέρει και τα αναγκαία εργαλεία για τις αγορές για να κάνουν τη μετάβαση αυτή προς ένα βιώσιμο μέλλον. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν πράγματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και να παραμένουμε ρεαλιστές. Γιατί τον κανονισμό αυτό θεωρώ ότι έχει μια πρόσθετη αξία και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι δεν είναι βιώσιμο. Όμως δεν είμαι πεπισμένοι ότι αν καθίσουμε να ελέγξουμε το κάθε επενδυτικό προϊόν για το κατά πόσο είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο, είναι κάτι που δεν προσφέρει η αναλογία, είναι δυσανάλογο με το κέρδος. Εγώ λοιπόν λέω ναι ε, για το, την πρόταση της Επιτροπής, όχι όμως για αυτήν ε, την αναλογική αντιμετώπιση για το τι είναι βιώσιμο και τι δεν είναι. Εγώ στηρίζω τον κύκλο ζωής ως προσέγγιση και χαίρομαι που πολλοί από εσά συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχής, καταρχάς να ευχαριστήσω τους συνηγητές, την ε, κυρία Πιέτη Κάινεν και τον κύριο Κάουτ, γιατί νομίζω ότι έχουν κάνει μια καλή δουλειά και έχουν εργαστεί παρά το ότι είναι γνωστό ότι έχουν και διαφορές μεταξύ τους να βρουν μια ισχυρή βάση συνένεσης για αυτόν τον τόσο σημαντικό ε, φάκελο, γιατί χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πλαίσιο και πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες είναι όχι να αποδυναμώνει, αλλά να ενισχύει όλα τα καλά στοιχεία που έχει η αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν. Με αυτό το πνεύμα χαρακτηρίζονται και οι τροπολογίες που κατέθεσα εκ μέρου της ε, ευρωομάδα τη Αριστεράς. Να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση του φακέλου, να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική, τη διάσταση περιβαλλοντικής προστασίας του φακέλου και να εγγυηθούμε μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, διαφάνεια και δίκαιη κατανομή των επενδύσεων. Θέλω να πω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί κινούνται γενικά σε μια θετική κατά τη γνώμη μου κατεύθυνση ε, και οφείλουμε να αντανακλούμε μέσα από αυτές μια πιο ισχυρή και πιο αποφασιστική προσέγγιση που οφείλει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο όνομα των πολιτών που μας εξέλεξαν. Αν δείτε το Ευρωβαρόμετρο η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει ισχυρότερες πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό είναι cross-party, είναι σε μια οριζόντια πολιτική βάση. Θα ήθελα μέσα από τις τροπολογίες που έχω καταθέσει να ενισχύσουμε κάποιες διαστάσεις. Πρώτον, να έχουμε μια πιο ρητή αυτοκριτική αναφορά σε αρνητικές εμπειρίες, όχι σε best practices, αλλά σε κακές πρακτικές, σε παθογένειες του παρελθόντος, όπου χρηματοδοτήσαμε λάθος πολιτικές ε, με ε, χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και αντίστοιχα, σε αντίστοιξη, σε κοντράστ με αυτό, να ε, ενισχύσουμε τα κριτήρια της αηφορίας και της ταξινόμησης αναδεικνύοντας ως, κριτήρια για τις βιώσιμες επενδύσεις. Ειδικά νομίζω ότι θα πρέπει να νοιαστούμε παραπάνω και για τους στόχους της μείωσης των ανισοτήτων, των διακρίσεων, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και θα ήθελα να υπογραμμίσω προς τους συνεισηγητές την τροπολογία 496 που έχω καταθέσει, θα ήθελα να τη δουν με ένα πιο ανοιχτό πνεύμα. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει σε όλο το κείμενο να αντανακλάται ισχυρά ο σεβασμός που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις κατευθυντήριε αρχές του ΟΗΕ. Διαπιστώνω ότι οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει η Ευρωομάδα τη Αριστερά, οι σοσιαλιστέ και οι Πράσινοι κινούνται σε πολύ σημαντικό βαθμό στην ίδια κατεύθυνση και γνωρίζω ότι η κυρία Πιετικάινεν είναι αρκετά ανοιχτή σε ε, τέτοιες προτάσεις που ενισχύουν και δεν αποδυναμώνουν τις βασικές κατευθύνσεις του φακέλου. Άρα θα ήθελα ένα-δυο βήματα παραπάνω σε αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι η τελική συζήτηση θα μας επιτρέψει και με τις ψηφοφορίες να πετύχουμε μια ευρύτατη συνένεση σε μια πρόταση που θα βελτιώνει και δεν θα αποδυναμώνει την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο παρακαλώ. Η κυρία Μπερές. Ναι, είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι καλό που μπορούμε να μιλήσουμε μετά τους σκιώδεις συζήτητες. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή. Αυτό που με θλίβει κάπως είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ο κανονισμός αυτός της ταξινόμησης ε, θα είναι κάπως χωριστός από τα άλλα ζητήματα. Αλλά χαίρομαι που με τις προτάσεις των συνεισηγητών μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μακριά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λάβουμε υπόψη μας την κυκλική οικονομία, τα απόβλητα, ε, τη σπατάλη και την διατήρηση, την προστασία της βιοπικιλότητας που είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση κυρίως για το θαλάσσιο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό όσο γίνεται πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί κατάλληλα για να αποφύγει αυτό που λέμε greenwashing. Δηλαδή ε, να έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα αναπτύσσει τη δικιά του στρατηγική αντί να μπαίνει στην στρατηγική που, για την οποία μίλησαν οι ειδικοί παγκοσμίω που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τα βιώσιμα οικονομικά. Ανοίγει λοιπόν μια συζήτηση για το τι θα συμπεριλάβουμε και τι όχι. Και οι εμπειρογνώμονε υψηλού επίπεδου το συζήτησαν για το αν πρέπει να έχουμε κριτήρια διακυβέρνηση και κοινωνικά κριτήρια. Εγώ θέλω να προσέξουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία, για παράδειγμα, ε, οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Αυτό όμως που κινητοποίησε την όλη διαμαρτυρία είναι η φορολόγηση των ε, καυσίμων. Και όλοι γνωρίζουμε ε, στην χώρα αυτή, στη Γαλλία, ότι μπορεί να συνάδει με τον οικολογικό φόρο, αλλά αναγκαστήκαμε να παρετηθούμε. Αν λοιπόν δεν λάβουμε υπόψη μας και τον κοινωνικό παράγοντα, θα την πατήσουμε. Παρόλο που θέλουμε να προωθήσουμε περιβαλλοντικούς στόχους, δεν το λέω αυτό μόνο επειδή είμαι ε, από του σοσιαλιστές και πάντα με ενδιαφέρουν τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά το λέω για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην προστασία του περιβάλλοντο. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και αυτά. Και ένα παράδειγμα έξω από την ταξινόμηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο καλύτερο τρόπο, εντάξει, ορισμένου δεν αρέσει, αλλά όπω εγώ πολλοί πιστεύουν ότι για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε φορολόγηση στον άνθρακα. Ναι, αλλά είναι αδύνατον αν δεν λάβουμε υπόψη μας την κοινωνική διάσταση. Και γι' αυτό θα ήθελα οι συνεισηγητές να είναι πολύ προσεκτικοί. Και μάλιστα το όφελος από την ταξινόμηση είναι ακριβώς ότι δεν χρησιμοποιούμε το εργαλείο της φορολόγησης που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για τους λόγους που σας εξήγησα, αλλά χρησιμοποιούν τον προσανατολισμό ε, προς τις επενδύσεις. Λαμβάνουμε υπόψη μας δηλαδή τις επενδύσεις και φτιάχνουμε ένα δίδυμο ε, περιβάλλον, επενδύσεις και από την άλλη μεριά κοινωνική διάσταση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να πετύχουμε. Ξέρω ότι πολλοί λένε και από την ομάδα εργασίας ε, των εμπειρογνωμόνων λένε «Μα προσοχή, μη βιαζόμαστε, ναι, αλλά θέλουμε συνοχή και αποτελεσματικότητα. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ευχαριστούμε. Άλλος. Όχι. Τότε θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Σπόλτς. Ο κύριος Σπόλτς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε καλοδεχόμενη εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό το επίγον θέμα και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές για τη σκληρή τους δουλειά. Σημειώσαμε τις ε, προτινόμενες ε, τροπολογίες ε, και το επίπεδο φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θεωρούμε ότι το πνεύμα των περισσότερων τροπολογιών πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά έχουμε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, για την ε, κατάταξη αυτή. Όπως ξέρετε, η προσέγγιση της Κομισιόν είναι ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τη μετάβαση της οικονομίας προς τα εκεί όπου θέλουμε. Έτσι, οι βιώσιμοι χρηματοοικονομικοί θα πρέπει να στηρίζουν τον ε, τομέα που ρηπαίνει αντί να τον τιμωρεί. Ε, αν λοιπόν επιμένουμε να κάνουμε κάτι στον τομέα αυτής της ε, νόμισης. Ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά του τι σημαίνει αυτό για τον τομέα της ε, ρευστότητας του να δημιουργήσουμε κάποια στοιχεία αποκλεισμένα, τρόποντινά και τον κοινωνικό αντίκτυπο επίσης τους πολίτες. Οπότε καλό θα ήταν να επιμείνουμε στην προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει, την πιο θετική να στηρίζουμε αντί να τιμωρούμε. Επίσης ε, είμαστε και επικεφαλής της ε, ομάδας ε, των ειδικών για την πράσινη ταξινόμηση. Η δουλειά προχωράει πάρα πολύ καλά, οπότε το να κάνουμε κάτι τώρα στον τομέα της καφέ της λεγόμενης ταξινόμησης απλά θα προσθέσει πολυπλοκότητα. Επίσης Είδαμε κάποιες ε, τροπολογίες που έχουν στόχο να προσθέσουν έναν επιπρόσθετο κοινωνικό στόχο. Προφανώς ε, θέλουμε να εργαστούμε για θετικά κοινωνικά αποτελέσματα στο γενικότερο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Ξέρετε ότι καλύπτεται εδώ πέρα η κοινωνική βιωσιμότητα σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάνει και μία πρόταση που καλύπτει την κοινωνική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της ε, νομοθετικής πρότασης για την αποκάλυψη. Επίσης έχουν εισαχθεί κάποιες ρήτρε σχετικές, αλλά αυτήν την στιγμή δεν πιστεύουμε απαραίτητος ότι η πρόσθεση επιπλέον στόχων ε, στον κανονισμό αυτόν θα έχει θετικά αποτελέσματα. Τέλος, ε, για τις κοινωνικές αυτές ρήτρε υπάρχει ήδη το άρθρο που έχει ακριβώς τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ε, όταν γίνεται αυτή η ταξινόμηση των περιβαλλοντικών στόχων και έχουμε ακριβώς ε, δεχτεί και κάποιες σχετικές Στη συζήτηση στο Συμβούλιο επίση τα πράγματα πηγαίνουν προ την ίδια κατεύθυνση, οπότε η Κομισιόν είναι ανοιχτή προ συζήτηση για να δούμε πώ θα ενισχύσουμε περαιτέρω αυτέ τι ε, ρήτρε για να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο συνομοθέτε. Αναμένουμε την συνέχεια των διαπραγματεύσεων και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στους ηγητέ. Ο κ. Σάιχαουτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω η συζήτηση αυτή δείχνει πως πράγματι γνωρίζουμε τα θέματα που συζητάμε και θα δούμε όπως είπαμε ειδικά την κοινωνική διάσταση γιατί ο στόχος των συνεισηγητών είναι να υπάρξει μια ευρεία πλειοψηφία για να έχουμε ακριβώς μια ισχυρή θέση στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο και θα πρέπει να εργαστούμε στις κοινωνικές πτυχές της ταξινόμησης αυτής για να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε έναν συμβασμό και το άλλο αφορά το πεδίο εφαρμογή. Ε, να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν όταν λέει ότι κάποιες από τις προτάσεις θα, μπορούσαν να θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ρευστότητα. Ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε να προλάβουμε είναι ότι οι επενδυτές μακροπρόθεσμα θα μείνουν με κάποια αποκλεισμένα στοιχεία ενεργητικού, προειδοποιούν οι εθνικές τράπεζες τότε θα υποστούν βλάβη οι επενδυτές. Πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι επενδυτές όταν έχουν μείνει με κάποια τέτοια στοιχεία στο χέρι τρόπον την Οπότε εμείς ε, ε, δεν ανησυχούμε μόνο για την ε, ρευστότητα την αυριανή αλλά και την μεθαυριανή. Πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη για να προετοιμάσουμε τον ε, χρηματοοικονομικό κλάδο να προετοιμαστεί για το μέλλον, όχι μόνο για το αυριανό αλλά και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ κυρία Πιατικάινεν. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επικοδομητικά της σχόλια και για τη δουλειά που έκανε προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε, να δίνουν πληροφορίες επενδυτές προς επιλογή αντί να δημιουργούμε ταξινομήσεις διαφόρων χρωμάτων. Αυτό δεν θα ήταν ε, πολύ επωφελές να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τα κοινωνικά θέματα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνώ με την Περβάνς Περές. Δεν μπορείς να κάνεις περιβαλλοντικές επιλογές και αλλαγές με κοινωνικό κόστος εις βάρος του λαού διότι δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα για μια κοινωνική ταξινόμηση ή λεπτομερέστατη προσέγγιση. Ας βρούμε κάποιο συμβιβασμό, τον οποίο μπορούμε να δεχτούμε όλοι, παρόλο που ίσως να μην είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι όλοι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους σας. Πολύ καλή συζήτηση επί των τροπολογιών. Προβλέπεται η κοινή ψηφοφορία των Επιτροπών 20 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Μάρτιο η ψηφοφορία. Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε. Εδώ ολοκληρώσαμε την κοινή συνεδρίαση. Και καλό τα μέλη περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος να πάνε στην αίθουσά μας για να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα σημεία της σημερινής διατάξής μας.